Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος. Ε, ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση και επί των ψηφισμάτων θα λάβει χώρα η ψηφοφορία αύριο στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε τώρα μία ανακοίνωση από τις ομάδες ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Άλντε και Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Έχω λάβει αιτήματα για ε, νέες θέσεις στις Επιτροπές ε, και τις αντιπροσωπή, κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες. Υπάρχει κατάλογος των εν λόγω ονομάτων. Εάν καμία παρατήρηση δεν θα έχει υποβληθεί μέχρι την έγκριση των πρακτικών, τότε αυτές οι νέες θέσεις θα των βουλευτών θα θεωρηθούν